κύριε πρόεδρε όταν περάσει να μπορούμε ο ένας να κοιτάζει τον άλλον. ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, σας ευχαριστώ για τις ομιλίες σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Επίτροπο που έμεινε μέχρι τέλος τη συζήτηση. Ε, ευχαριστώ και τους συνεργάτες μας ε, και τους διερμηνείς που υπερέβησαν και το ωράριό τους και να σας ανακοινώσω ότι θα συνεχίσουμε αύριο ημέρα 5η 2 Φεβρουαρίου στις 9 μέχρι τις 2. Το πρόγραμμα το έχετε. Υπάρχει και στην ιστοσελίδα. Διακοπή της Συνόδου. Καλό σας βράδυ.